και θα περάσουμε στο επόμενο σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη που αφορά στην έκθεση της κυρίας Εσάγια με θέμα ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Και θέλω πρώτα απ' όλα να παρακαλέσω την ε, εισηγήτρια, την κυρία για τέσσερα λεπτά. Κυρία Εσάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Είναι ένα πολύ τεχνικό θέμα αυτό. Είναι μια πολύ τεχνική έκθεση και ευχαριστώ τους κοιόδης εισηγητές για την καλή συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ τους βοηθούς μου επίσης και την Επιτροπή για την πραγματογνωμοσύνη της και για τον τριμερή διάλογο που οργάνωσε. Λοιπόν, περί τίνος πρόκειται. Είναι ένα θέμα ετικετοθεσίας και συσκευασίας που βασίζεται στους σχετικούς κανονισμούς. Μιλάμε για ένα σύστημα του ΟΗΕ για την αναγνώριση και την επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών για τους καταναλωτές. Με βάση το σημερινό σύστημα, οι κίνδυνοι των χημικών ουσιών γνωστοποιούνται στους καταναλωτές μέσω συγκεκριμένη διατύπωση και μέσω τη επισήμανσης. Μέσω τη αντικειτοθεσία δηλαδή. Έτσι ενημερώνονται. Όταν υιοθετήθηκε ο κανονισμός, καταλάβαμε ότι έπρεπε να γίνουν κάποιες τεχνικές προσαρμογές. Γιατί υπάρχει μία αναφορά στην Ευρωπαϊκή ε, Νομοθεσία για την επισήμαση των χημικών. Όλες οι αλλαγές έχουν να κάνουν με τέτοιου είδους τεχνικές ε, αναφορές, με αυτά τα τεχνικά σημεία. Αυτή η αναφορά στις πέντε σχετικές οδηγίες και η προσαρμογή της ε, διατύπωσης δεν απαιτεί καμία αλλαγή του πεδίου εφαρμογή των οδηγιών. Ούτε αλλάζει καθόλου το επίπεδο της προστασίας. Μπορούμε λοιπόν να προβούμε σε αυτή την αλλαγή, σε αυτή την τεχνική προσαρμογή. Όλα αυτά που λέει το επεξηγηματικό σημείωμα νομίζω είναι πολύ σημαντικά, γιατί στο μεταξύ υπήρξαν τεχνολογικές εξελίξεις και αυτές οι πέντε οδηγίες θα πρέπει να αναθεωρηθούν και ούτως ή άλλως να αναθεωρούνται και σε τακτή βάση για να προσαρμόζεται η νομοθεσία στις τεχνολογικές εξελίξεις για να εξασφαλίσουμε και το σωστό επίπεδο προστασίας όταν έχουμε να κάνουμε με τις χημικές ουσίες και τα μείγματα στο χώρο εργασίας. Επίσης, να σας επιστήσουμε την προσοχή σε κάποια επαγγέλματα και τους εργαζόμενους φυσικά σε αυτά τα επαγγέλματα που σε καθημερινή βάση έρχονται αντιμέτωποι με αυτές τις χημικές ουσίες και τα μείγματα και συχνά χωρίς την απαραίτητη προστασία. Χρειάζεται ειδική προστασία για αυτούς τους εργαζόμενους σε συγκεκριμένους κλάδους και, και γίνεται σχετική αναφορά σε μία τροπολογία. Επίσης, μιλάμε για τις εγγύους και τις θυλάζουσες μητέρες που εργάζονται σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Το ίδιο ευάλωτη μπορεί να είναι και οι νέοι, γιατί μπορεί να αντιδρούν σε κάποια περοξίδια, σε κάποιες πτυτικές ουσίες, σε κάποιες επικίνδυνες ουσίες. Θα θέλαμε λοιπόν να υπάρξει και σχετική αναφορά και στους νέους και στην ανάγκη για προστασία τους. Η προστασία στον χώρο εργασίας δεν θα αποτελέσει πρόβλημα. Χάρη σε αυτό το νομοθετικό μέσο και στην προστασία του Κοινοβουλίου υπάρχει ευρή αποδοχή. Είναι πολύ σημαντικό στο μεταξύ βέβαια να μην επιβαρύνουμε περιτά με περί τη γραφειοκρατία της μικρομεσαίας επιχειρήσης. Τούτου λεχθέντους βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε και το μέλημα για προστασία. Των εργαζομένων. Η προστασία των εργαζομένων δεν πρέπει να θεωρείται ποτέ βάρος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις εταιρείες, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Ο Επίτροπος, ο κύριος Άντορ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλω να εκφράσω τη χαρά μου για την ευκαιρία που δίνεται να συζητήσουμε την οδηγία αυτή. Η πρόταση οδηγίας είναι ένα ξέρετε έργο σε κάθε επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, τρεφύτερη εκτίμηση για τις ε, συμβολές των θεσμικών οργάνων και πιστεύει ότι το τελικό κείμενο ορίζει ικανοποιητικούς στόχους κοινού για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων στην Ευρώπη. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση που εξασφάλισε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο και ε, που προχώρησε σε στενή συνεργασία από πλευρά τη εισηγήτρια εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την αντίστοιχη ομάδα του Συμβουλίου, οδηγεί σε ένα κοινό κείμενο που στόχο έχει την συνέχιση της προστασίας σε υψηλό επίπεδο των εργαζομένων από πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με την έκθεση σε χημικές ουσίες στον χώρο εργασίας. Οι βελτιώσει σε σχέση με την πρόταση, όπως συμφωνήθηκαν στις διαπραγματεύσει, καταλήγουν σε ένα κείμενο το οποίο είναι όχι μόνο σαφέστερο νομοτεχνικά, αλλά και πιο εύληπτο. Και έτσι μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη υλοποίηση, μεταφορά και υλοποίηση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας και ως εκ τούτου βελτιώνω την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων. Συνεπάγεται δε την εισαγωγή ενό νέου συστήματο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση των ε, και επισήμανση των χημικών ουσιών, με μια πρόταση που υιοθετήθηκε το 2008 και προοδευτικά τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο σύστημα λοιπόν το οποίο εφαρμόζει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ε, παγκόσμιο και εναρμονισμένο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την ταξινόμηση και την επίσημαση χημικών προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών. Αναφέρεται εδώ όχι μόνο στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά κάνει και μια γενικότερη συμβολή, προσφέρει και μια γενικότερη συμβολή ως προς την ε, ε, ορολογία και την νομοθεσία. Και έτσι εξασφαλίζει καλύτερη αντίληψη για θέματα διαχείρισης κινδύνου μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όχι μόνο και με τους κύριους εμπορικούς μας εταίρους ανά τον κόσμο. Έχουμε λοιπόν δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ένα ευρύ φάσμα υλικού που μπορεί να, μπορεί να προσφέρει κατευθυντηρίες γραμμές, χρήσιμο και για τους ε, ε, για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τη λειτουργία του νέου συστήματος. Ε, καθοδήγηση λοιπόν την οποία προσφέρει δωρεάν ο Ιστότοπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθοδήγηση η οποία προκύπτει κατόπιν ε, διαβουλεύσεων με τους ε, φορείς. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους των πολιτικών ομάδων ξεκινάμε με τον κύριο Κρίστενσεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ τον εισηγητή για το πνεύμα συνεργασία που έδειξε. Είναι σημαντική πρωτοβουλία αυτή για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών από παλιά. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να εργάζεται σε συνθήκες που θα επινοούν την ασφάλεια και την υγεία του. Τέτοιου είδου μέτρα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ε, ως γραφειοκρατία. Η, η Κομισιόν ε, δεν έχει καταφέρει να δει το θέμα αυτό και από τις δύο μεριές με ισορροπία. Το να λέει ότι ο καθένας μπορεί να τα βγάλει πέρα μόνος του δεν είναι σωστό ε, και δεν είναι σωστή αυτή η προσέγγιση της Κομισιόν στην, στο πλαίσιο ενός κοινωνικού διαλόγου. Θα πρέπει η Κομισιόν να αναλάβει τις ευθύνες της σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό διάλογο με τους εταίρους. Έχω εργαστεί επί μακρόν σε θέματα επισήμανσης και συσκευασία. Πιστεύω ότι τέτοιου είδου προδιαγραφές και πρότυπα δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως άχθος. Δεν θα πρέπει να, να μετράτε μόνο το κόστος τους. Και δεν θα πρέπει το κόστος να, θεωρεί, να χρησιμοποιείται ως αφορμή για να ε, μην αναλάβουμε δράση. Πρέπει να αποφύγουμε τα, τους τραυματισμούς στον χώρο εργασίας, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επικίνδυνες χημικές ουσίες. Πρέπει να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στη βιομηχανία, στα εργοστάσια, ε, ακόμα και στα κομμωτήρια. Στα κομμωτήρια, για παράδειγμα, εκτίθενται σε πολλές χημικές ουσίες, ε, τις οποίες, των οποίων τους κινδύνους πολλές φορές δεν γνωρίζουμε. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Η, συνάδελφος Χάρκιν, Μαριάν Χάρκιν. Thank you. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, την εισηγήτρια για τη ρεαλιστική προσέγγιση που έχει σε αυτό το νομοθέτημα. Πρέπει να ενισχύσουμε τον κανονισμό της ε, υγείας και την ασφαλειας για τους εργαζόμενους. Υπάρχει ένα αρμοσμένο σύστημα για την ταξινόμηση των χημικών του ΟΗΕ, το 2005 υιοθετήθηκε και είναι σημαντικό για την ασφαλεία και την υγεία των εργαζομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε πέντε οδηγίες για την υγεία και την ασφάλεια που χρησιμοποιούν τις παλιές αναφορές στην παλιά ταξινόμηση και στο παλιό σύστημα ταξινόμησης. Χρειάζεται λοιπόν ευθυγράμμισή τους με τη νέα νομοθεσία. Και αυτό γίνεται. Έχουμε επικαιροποίησει τις αναφορές, την ορολογία, ούτως ώστε να απεικονίζεται και να παραπέμπουμε στο νέο σύστημα που χρησιμοποιούμε. Συμφωνώ με τον κατάλογο των ευπαθών εργαζομένων που έχουμε προσθέσει, τους νέους, τις εγγύους κτλ. Και συμφωνώ επίσης με τις συστάσεις ότι επεξηγηματικές κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να δοθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, δεν πρόκειται για επιπλέον υποχρεώσεις και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως επιπλέον ναύτος για τις επιχειρήσεις αυτές οι ανάγκες για προστασία των εργαζομένων και για ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι σημαντικό να νομοθετούμε υπέρ τη ασφάλεια και τη υγεία των εργαζομένων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση να επενδύσουμε προκειμένου να προλάβουμε τραυματισμού και ατυχήματα στο χώρο εργασία σε σχέση με τι επικίνδυνε χημικέ ουσίε. Υπάρχουν πέντε σχετικέ οδηγίε με ε, ελάχιστε προδιαγραφέ για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία. Η οδηγία την οποία συζητούμε διατηρεί ένα επίπεδο προστασία των εργαζομένων ε, που ήδη η πρόταση του Κοινοβουλίου υπογραμμίζει ότι ε, δεν θα πρέπει να βλέπουμε το θέμα περιοριστικά. Πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θα πρέπει να μπορούν να ασκηθούν χωρίς περιορισμού σε όλα τα περιβάλλοντα εργασία και σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Συμφωνούμε, όλα αυτά είναι σωστά και επιθυμητά. Δυστυχώς όμως όταν δούμε, βλέποντας την πραγματικότητα, αυτή διαφέρει από τη θεωρία και από τον νόμο. Είναι γνωστό ότι τα ατυχήματα λαμβάνουν χώρα σε άμεση συνάρτηση με την επισφάλεια στο χώρο, των θέσεων εργασία. έχουν σχέση επίσης ε, με την αδυναμία οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και με την έλλειψη κατάρτισης και επένδυσης επενδύσεων σε θέματα πρόληψης. Οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται υπό οποιασδήποτε συνθήκες πλέον και οι συνθήκες εργασίας ε, έχουν χειροτερέψει σε σχέση με το παρελθόν. Ε, χρειάζεται έλεγχος, χρειάζεται δημόσια επένδυση, χρειάζονται εγγύησεις και χρειάζεται να εξασφαλίσουμε τα θέμα, ε, και χρειάζεται εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια. Ε, μόνο έτσι θα αποφύγουμε τα ατυχήματα. Επίσης χρειάζεται να προβλέψουμε επαρκείς επανορθώσεις ε, σε περίπτωση ατυχημάτων. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει πολλά ε, ατυχήματα ε, τέτοιου τύπου, ιδιαίτερα στις χώρες οι οποίες υποστηρίζονται από το Διεθνές Μεσονοτικό Ταμείο. Και πρώτα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο για την καλή της έκθεση και για όλες τις προσπάθειες που έχει αναπτύξει. Είναι πολύ σημαντικό να προστατέψουμε την υγεία στο χώρο εργασίας και χαίρομαι που έχουμε παρόντα τον Επίτροπο Άντορ γιατί ίσως θα μπορούσε να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις ως προς τις έρευνες στα επαγγελματικά νοσήματα στην γεωργία που προκαλούνται από την έκθεση σε γεωφαρμακευτικά προϊόντα. Ευχαριστώ. Αυτή η οδηγία πραγματικά καθορίζει τι είναι προστασία των εργαζομένων. Χρειάζεται να προστατεύουμε ιδιαίτερα αυτούς που υφίστανται κινδύνους εξαιτία χημικών ουσιών. Αυτό δεν αποτελεί άκθος και γραφειοκρατία. Ο κατάλογος των ε, επαγγελμάτων ε, θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο κοινωνικός διάλογος θα είναι το μέσο προκειμένου να εφαρμόζονται τέτοιου είδους οδηγίες. Είναι αλήθεια ότι τέτοια νομοθεσία συνήθως επηρεάζει εργαζομένους που υφίστανται σημαντικούς κινδύνους και προβλήματα, για παράδειγμα στην κλωστοεφαντουργία. Και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και εγώ, η συνάδελφος Μπασέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μπορεί να συστούμε μια πρόταση που έχει τεχνικά χαρακτηριστικά, ε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία η έγκρισή της για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του χώρο εργασίας, ε, για τη συσκευασία των ουσιών και την επισήμανσή τους. Ε, ως μικρομάνα θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνεται αναφορά και να είναι ενήμερος ο για τις ουσίες τοξικές, καρκινογόνες και άλλες ε, διότι μπορεί κατά την εγκυμοσύνη να προκληθεί ζημιά και στο έμβριο ακόμη και έτσι να γεννηθεί το μωρό άρρωστο και μητέρες που θυλάζουν κινδυνεύουν να μεταδώσουν κάποια νοσήματα στο παιδί τους και καθώς το ανασωπητικό του παιδιού δεν είναι ε, αρκετά ε, εξελιγμένα, είναι πολύ πιο εκτεθειμένα τα νεογέννητα και τα βρέφη στην ε, έκθεση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία. Ευχαριστώ, Επίτροπο Σαντόρ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και τα στοιχεία προβληματισμού που δίνεται στην Κομισιόν, η Κομισιόν περιμένει τώρα την υιοθέτηση της πρότασης από το Συμβούλιο και τη δημοσίευση της οδηγίας στην επίσημη εφημερίδα. Είμαι πεπισμένος ότι είναι μια σημαντική συμβολή στην προστασία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο, στους χώρους εργασίας τους. Όπως είπε και ο κ. Κρίστιανσεν, ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι πολύ σημαντικό, ήταν και είναι. Κύριε Νικολέσκου, να σας πω ότι παρότι είναι σημαντικό να τονίσουμε το ρόλο ορισμένων τομέων, το βασικό μας θέμα στην νομοθεσία είναι πώς αντιμετωπίζουμε συγκεκριμένους κινδύνους μέσα από ένα νομοθέτημα σε διάφορους οικονομικούς τομείς. Παραδείγματο χάρη στην έκθεση στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η απάντηση είτε είναι ο α ή ο β κλάδος, ε, πρέπει να είναι η απάντηση η ίδια. Κυρία Χάρκιν, ε, εστιάζουμε ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφωθούν με την νομοθεσία χωρίς να τις επιβαρύνουμε υπερβολικά όμως. Όλα όσα άκουσε η Κομισιόν θα βοηθήσουν περαιτέρω την Κομισιόν στο να προωθήσει αυτά τα νομοθετήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαϊά, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούσαμε στην συζήτηση ότι παρόλο ότι διαθέτουμε πολύ λεπτομερείς κανόνες για τις επικίνδυνες ουσίες, αυτοί οι κανόνες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως γραφειοκρατικοί. Είναι σημαντικοί για να εξασφαλίσουμε την υγεία και την ασφάλεια των αζωμένων. Χρειάζεται όμως όλες οι επιχειρήσεις να είναι ενήμερες, ιδιαίτερω μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, ε, γι' αυτό το λόγο έχει δίκιο ο κύριος Σάντορ. Στην Κομισιόν υπάρχει ήδη μια σελίδα όπου ένας επιχειρηματίας μικρομεσαίας επιχείρησης μπορεί δωρεάν να πάει και να βρει πληροφορίες έτσι ώστε να είναι ενήμερος. Το λέμε και εμείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να μπορούν να ενημερώνονται. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ κυρία Εσάγια. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και θέλω να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30. Θα περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις διάρκειας ενός λεπτού και πρώτα θέλω να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Πρέντα.